Θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τους συντάκτες της ερώτησης, των ψηφισμάτων. Ε, ο κύριος Κέλαμ θα πάρει το λόγο πρώτος για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Το Ιράν είναι ε, περιβόητο για τις παραβιάσεις ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν συνέβη αυτό μόνο χθε. Σήμερα όμως ε, εξετάζουμε την περίπτωση της Ροξάνα Σαντζέρη, της δημοσιογράφου, της οποίας η δίκη έγινε μόλις πριν από τρεις εβδομάδες και καταδικάστηκε σε οκτώ χρόνια φυλάκιση για κατασκοπία. Είχε λοιπόν ε, η δυνατότητα να έρθει σε επαφή με το δικηγόρο για ένα μήνα περίπου, αλλά παρόλα αυτά δεν είχε δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, γιατί ήταν η δίκη και κλεισμένων των θυρών. Έτσι λοιπόν δίρκεσε η δίκη δύο εβδομάδες, μόλις ολοκληρώθηκε. Η υγεία της όμως ε, είναι ε, πλέον σε πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Έχουμε τη δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με ε, το επαναστατικό δικαστήριο του Ιράν ε, να αμφισβητήσουμε την απόφασή τους που εκδόθηκε στις 18 Απριλίου και πρέπει να ζητήσουμε, η κυρία Σαμπέρη, παρά αυτά και χωρίς όρους να αφηθεί ελεύθερη διότι όπως είπαμε η δίκη έγινε και κλεισμένων των θυρών χωρίς να τηρηθεί η ποινική οικονομία. Το Ιράν όλοι μας γνωρίζουμε ότι είναι περιβόητο ε, για τις εκτελέσεις που λαμβάνουν χώρα στην ε, πόλη, για τον απαχανισμό, τη δολοφονία, ε, ακόμα και ανηλίκων. Έτσι λοιπόν οι λιθοβολισμοί και οι επαγχωνισμοί είναι κάτι που το γνωρίζουν όλοι. Για λεπτό. Eh, eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα τελευταία πέντε χρόνια έγιναν πολλές συζητήσεις σχετικά με το Ιράν. Η ομάδα μου ήταν υπέρ της επανάστασης κατά το τέλος του δεκαετή, της δεκαετίας του 80 γιατί η οικογένεια Παχλεβή δεν εκπροσωπούσε τον λαό και αυτή η κυβέρνηση είχε επιβιώσει εξαιτία των δεσμών με την Αμερική τότε. Όμως, στην αρχή της Επανάστασης είδαμε ότι η κατάσταση ήταν διαφορετική και οι πολίτες τράφηκαν κατά της δύση. Οι Δυτικοί θεωρήθηκαν μία απεικιοκρατική δύναμη εκμετάλλευσης. Τώρα βλέπουμε ότι έχουμε να κάνουμε με ακραία στοιχεία που τάσσονται κατά του Ισραήλ. Δεν υπάρχει πραγματική δικαιοδοσία και ο θρησκευτικός ε, φονταμενταλισμός οδήγησε σε μια ακραία στάση. Δεν υπάρχουν δικαιώματα για τις γυναίκες και η ποινή θανάτου πολλές φορές ε, γίνεται ενώπιον κοινού, κατά βάνουσο τρόπο. Επίσης, Κανένας δεν μπορεί να αντιταχθεί σε αυτή την κυβέρνηση. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε με μια κατάσταση, μια ακραία κατάσταση εθνικισμού και θα πρέπει η αντιπολίτευση, μάλλον η αντιπολίτευση ε, θεωρείται ως μια τρομοκρατική οργάνωση. Θεωρούνται ε, τρομοκράτες. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό που έχει σημασία είναι να λάβουμε υπόψη αυτή την κατάσταση βίας που ενδυνάμωσε το καθεστώς. Όλοι μισούν την παρούσα κυβέρνηση, αλλά υπεραμείνονται της χώρας. Κρατήσατε πολύ τον χρόνο. Ο κύριος Καζάκα είναι ο επόμενος ομιλητής. Κρατήστε το, τα δύο λεπτά. του minutes, Mr. Καζάκα, please. Η 1η Μαΐου που είναι η μέρα του εργάτη δυστυχώς είναι μία μέρα θλίψης για το Ιράν και πένθους για το Ιράν διότι έχουμε να κάνουμε με ε, εκδηλώσεις και διαδηλώσεις που οδήγησαν στο, στην ε, καταδίκη της διλάρα Νταράμπη η οποία ήταν 17 χρονών. Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, μία μέρα πριν από την εκτέλεση αυτής της νεαρής, η νεαρή αυτή, η Διλάρα Νταράμπη, είχε πει στη μητέρα της ότι θα ήθελε να απελευθερωθεί. Η Διλάρα Νταράμπη ήταν ε, απότοκο ενός ε, φανατισμού γενικότερα. Νομίζω λοιπόν ότι δεν μπόρεσε να υπάρξει επιβεβαίωση του λιθοβονισμού ενός ε, ανθρώπου στην, ε, στην φυλακή του Λάκεν. Και βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η βάρβαρη πρακτική συνεχίζεται, η πρακτική του λιθοβονισμού. Βλέπουμε λοιπόν ότι στο Ιράν υπάρχουν περισσότερες κατακεφαλή εκτελέσεις σε σχέση με όλες τις χώρες του κόσμου, διότι στο ΕΒΙΝ καταδικάστηκαν σε θανατική ποινή τέσσερις κρατούμενοι που είχαν ε, καταδικαστεί στις 2 Μαΐου. Και η Αμερικανή Ροξάνα Σαμπέρι ακολούθησε αυτή τη, τη ρουτίνα δυστυχώς την καταδίκη της. Αυτό που έχει σημασία είναι η δήλωση του Σέργιο Ντέλια. Οι μουλάδες ε, ακολουθούν μια εκφοβιστική πολιτική, μια βάναυση πολιτική, χωρίς να υπάρχει ανεκτικότητα και υποκύπτοντας στον εκβιασμό της ε, πολιτικής του Ιράν. Πιστεύω λοιπόν ότι το καθεστώς του Τεχεράν διαιωνίζει αυτή την κατάσταση εκφοβισμού των πολιτών τους. Εφόσον μιλώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τελευταία φορά, εύχομαι αυτοί που θα ασχοληθούν στην επόμενη θητεία να μην εγκαταλείψουν τους Ιρανούς κατά την επόμενη θητεία σε αυτό τον ε, φανατισμό, θρησκευτικό φανατισμό. <clears throat> Σας έκανα και δώρο λίγα δευτερόλεπτα, επειδή είναι η τελευταία φορά που μιλάτε. Ε, τώρα ο κύριος Ματσάκης, συντάκτης επίσης, για δύο λεπτά. Madam President, I will not repeat what... Κύριε Πρόεδρε, δεν θα επαναλάβω αυτά που έχουν ήδη ληχθεί όσον αφορά ε, το ε, αδίστακτο Ιρανικό καθεστώ. Συμφωνώ με όλα αυτά. Εγώ όμω θέλω να εξετάσω το θέμα κάτω από ένα άλλο πρίσμα από αυτό ε, το οποίο παρουσίασε ο κύριο Μάγερο, συνάλφο που μόλι έφυγε. Το Ιράν έχει χιλιάδε έτη πολιτισμού και ιστορία. Σήμερα βρίσκεται σε μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση όσον αφορά τη δημοκρατία και τα κοινωνικά δικαιώματα. Ορισμένε χώρε στη Δύση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 καταδικάζουν ε, αυτή την κατάσταση. Οι κυβερνήσει όπω οι ΗΠΑ και η Μεγάλη Βρετανία για, χίλια, για ολόκληρα χρόνια βοήθησαν το Ιράν, έδιδαν όπλα στο, ε, στη δικτατορία του Σάχη στο Ιράν. Ήταν λοιπόν αναπόφευκτο όταν πλέον ανετράπη ο Σάχη από κοινωνική αναταραχή, οι Ισλαμιστέ, ε, ακραίοι εθνικιστέ και φανατικοί θρησκευόμενοι θα έβρισκαν πρόσφορο έδαφο για να καλλιεργήσουν το μίσο ει βάρο τη Δύση. Κατόπιν ακολούθησαν οι ε, ε, επιβολή κυρώσεων που και αυτό προκάλεσε επίσης ε, πόνο στους Ιρανούς και όξινε τα αρνητικά τους και εχθρικά τους συναισθήματα προς τη Δύση. Ευχόμεθα ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κύριος Ομπάμα, που δείχνει ότι θέλει περισσότερο να αγωνιστεί με το μυαλό του και όχι με την πυγμή του, όπως το έκανε ο προκάτοχός του. Ας ελπίσουμε ότι ο νέος πρόεδρος θα δώσει νέα βάση ελπίδες για βελτίωση των σχέσεων με τη Δύση. Μια τέτοια στάση θα βοηθήσει του Ιρανού να κατανοήσουν ότι η Δύση επιθυμεί να είναι φίλο του και όχι εχθρό του. Και με το χρόνο οι πολίτε του Ιράν μόνοι του θα ανατρέψουν το φονταμενταλιστικό αυτό καθεστώ, ε, το οποίο ε, αντιδημοκρατικά ελέγχει τη ζωή του και προκαλεί τόσο μεγάλο πόνο όπως στην περίπτωση αυτή που συζητάμε σήμερα και ε, θέλω να σας πω απίστευτο αλλά τέλειωσα και 10 δευτερόλεπτα πριν από το χρόνο που μου είχατε διαθέσει. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και οι συνάδελφοι, δεν θα καθυστερήσουμε. Ε, η κυρία Τομαζεύσκα για δύο λεπτά παρακαλώ. Πάνη Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Ροξάνα Σεβέρη, είναι δημοσιογράφο, 32 ετών. Έχει διπλή πηγότητα. Είναι απόφυτος διαφόρων πανεπιστημίων στις ΗΠΑ, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Ιράν. Ο δημοσιογράφος στο Ιράν καταδικάστηκε σε φυλάξη 8 ετών με πρόσχημα την τεχνητή κατηγορία της κατασκοπίας. Διαμαρτυρήθηκε βεβαίως για τις αστερικές κατηγορίες και ξεκίνησε περιγεπίνας. Αυτή τη στιγμή έχει σταματήσει την απεργία πείνας και αναμένει το αποτέλεσμα της έφεσης που έχει ασκήσει. Το Ιράν είναι διαβόητο για τις ε, δημόσιες εκτελέσεις που εφαρμόζει μεταξύ άλλων και ανηλίκων. Καλούμε το Ιράν να απελευθερώσει την κυρία Σαμπέρη και να της εξασφαλίσει δίκαιη δίκη οφείλουμε να πιέσουμε το Ιράν να σταματήσει αυτές τις απαραδείκτες πρακτικές. Εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων θα ξεκινήσουμε με την κυρία Ανδριεκένε για 1,5 λεπτό εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Έχετε το λόγο. Mes kalbame apie Amerikos Κύριε Πρόεδρε, μιλάμε για τον Ροξάνα Σεπέρι. Είναι δημοσιογράφο που έχει δουλέψει το ABC, το BBC και την νοτιοφρικανική τηλεόραση. Κατηγορήθηκε για κατασκοπία και καταδικάστηκε σε φυλάξη 8 ετών. Όπως γνωρίζετε, ξεκίνησε απεργία πείνα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο των φυλακών με την υγεία τη σε εξαιρετικά ευθαρστή κατάσταση. Δεν είχε πρόσβαση δικηγόρο για πέντε εβδομάδε. Η δίκη της διεξήχθη σε καθεστώς αδιαφάνεια. Αυτά τα ανακοίνωσε το BBC στις, τελευταίε τελευταίες εβδομάδες. Στις 12 Μαΐου το εφετείο θα ασχοληθεί με την εφησή τη, αλλά και πάλι η δίκη αυτή θα γίνει και κλεισμένα των θυρών. Καταδικάζουμε την αδικαιολογητή ποινή του επανθερικού δικαστηρίου κατά της ξανα Σαμπέρι. Καλούμε τις Ιρανικές αρχές να σεβαστούν τα διάφορα κείμενα για τα δικαιώματα του ανθρώπου και κυρίως τον Οικουμενικό Χάρτη. Και να εξασφαλίσουμε βεβαίω δίκαιη δίκη. Πάρει το λόγο εκ μέρους της ε, σοσιαλιστικής ομάδας. Ε, Κυρία Πρόεδρε, τελευταία μέρα σήμερα βεβαίω. Η άνοιξη δεν περνάει παρατήρητη. Θα ήταν πιο ευχάριστο εάν η σημερινή μας συζήτηση περί δεν είχε ούτε ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη. Δυστυχώ, η ημερήσια διάταξή μα είναι φορτωμένη. Και πάλι δεν έχουμε καταφέρει να συμπεριλάβουμε τι διάφορε υποθέσει που μα απασχολούν. Δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμε με το Ιράν. Αυτή τη φορά μιλούμε για την παράνομη φυλάξη τη Ροξένας Σαβέρη. Σε αρχή συνελήφθη για πλημέλημα μια κατοχή Ινούπ, το οποίο είναι παράνομο Μετά καταδικάστηκε διότι υποτίθεται ότι ρίζονταν χωρί την απαραίτητη άδεια και στο τέλο κατηγορήθηκε ότι δούλευε ω κατάσκοπο υπέρ των Αμερικανών. Αυτά κρίθηκαν κατά τη διάρκεια μια δίκη που δίρξε μόλι μία ημέρα χωρί να τι επαγγελθούν επισήμω κατηγορίε. Οι Ιρανικέ αρχέ, δεν υπάρχει καμία εμφιβολία, καταπατούν τα δικαιώματα του ανθρώπου. Γνωρίζουμε για την εκτέλεση τη Δελάρα Νταράμπη. Γνωρίζουμε για τη σύλληψη τη Μαριάν Λακμπή και άλλων δημοσιογράφων. Αυτή και αυτά είναι μόνο μερικά από τα παραδείγματα που γνωρίζουμε. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι τα ακραία στοιχεία, οι φανατικοί στο Ιράν, χρησιμοποιούν παράνομες δίκες για να καταπνίξουν την ελεύθερη σκέψη. Το Ιράν αυτοκομονώνεται και δεν σκοπεύει να συμμετάσχει στον διάλογο με την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα. Έχει επιλέξει την αντιπαράθεση. Προτείνω συναφώς να δώσουμε μια πολύ σκληρή απάντηση στην συγκεκριμένη αυτή περίπτωση. Να ζητήσουμε λοιπόν από το καθεστώς να γίνει κάνει σεβαστά τα δικαιώματα του ανθρώπου. Κρούπα, η οποία όμως δεν βρίσκεται στην αίθουσα και έτσι θα πάρει το λόγο ο κύριος Στέμψον για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε η φυλάκιση της Ροξάνα Σαμβέρη με την κατηγορία της κατασκοπίας ε, είναι ένα επονίδιστο γεγονός, άλλο ένα έγκλημα σε αυτό τον μακρύ κατάλογο καταχρήσεων ε, στις οποίες προβαίνει το φασιστικό καθεστώς στο Ιράν. Την περασμένη Παρασκευή, όπως μας είπε ο κύριος Καζάκας, την εξετέλεσαν, εξετέλεσαν ένα κορίτσι 23 ετών, ε, το πήραν από το κελί ε, και την εξετέλεσαν χωρίς να επιτρέψουν να τη δουν οι γονείς της. Ε, την κρέμασαν για εγκλήματα που αρνείτο. Υποτίθεται είχε κάνει έγκλημα στα 17 και το αρνείτο συνέχεια. Στο Ιράν υπάρχουν βασανιστήρια και εκτελέσεις εις βάρος γυναικών και παιδιών, ακόμα και εγγύων και αυτό είναι μια καθημερινή μακρινή πρακτική. Παρόλα αυτά έχουμε κυρία Πρόεδρε σε αυτό το κοινοβούλιο ανθρώπους οι οποίοι υποστηρίζουν αυτό το διεφθαρμένο και παράνομο καθεστώς. Ακριβώς όπως εκείνες οι ευρωπαϊκές εταιρείε που συνεχίζουν να συνδιαλέγονται οικονομικά με το Ιράν. Τα αυτιά τους και τα μάτια τους ε, έχουν κλείσει στις φωνές του τύπου. Ντροπή τους, <clears throat> ντροπή στους ε, βίαιους μουλάδες. Δεν πρέπει να ξεχνάνε τα μαθήματα της ιστορίας. Όλα τα φασιστικά γεγονότα είναι καταδικασμένα να αποτύχουν. Η ελευθερία και η δικαιοσύνη θα υπερισχύουν πάντα του κακού. Ο κύριος Μέγερ παρόλο το ότι είχε παρέμβει ε, θέλει να κάνει μια σύντομη τοποθέτηση. Σύντομα, όχι περισσότερο από ένα λεπτό κύριε Μέγερ σας παρακαλώ. Eh, Κυρία Πρόεδρε, Σωστά. Ε, μου κόψατε προηγουμένως ε, το λόγο γιατί ε, μίλησα παραπάνω. Μόνο που θέλω να πω ότι ε, η διεθνής παρέμβαση δεν βοηθάει σε τίποτα στο Ιράν. Φτάσαμε στην κατάσταση που φτάσαμε. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ε, μισούν την κυβέρνηση, όμως παρόλα αυτά θέλουν να υποστηρίξουν την πατρίδα τους. Είναι ε, λάθος να θέλει κανείς να συνεργαστεί με την κυβέρνηση απλά και μόνο για να υπάρχει σταθερότητα στην παροχή ενέργειας. Η στήριξη της δημοκρατικής αντιπολίτευσης είναι ο μόνος σωστός δρόμος, αυτός που θα έπρεπε να ακολουθεί και για το θύμα για το οποίο συζητάμε σήμερα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να στηρίξω τον συνάδελφό μου, τον κύριο Στίβενσον, ακόμα και να είναι Σκοτσέζος. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η Περσία, ο Περσικός ήταν ένας από τους μεγαλύτερους πολιτισμούς σε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχουν πολλοί Ιρανοί που είναι αξιοπρεπείς και σοβαροί άνθρωποι. Ο Στίβεν μίλησε από την καρδιά του και έχει δίκιο. Κανένας άνδρας δεν μπορεί να σκοτώνει ε, γυναίκες ε, και παιδιά και να επέρεται γι' αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε. Εμείς ε, είμαστε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να φωνάξουμε, να ε, δώσουμε έκφραση στην οργή μας ε, κατά αυτής της απάνθρωπης συμπεριφορά. Και εγώ καταλήγω στο ότι πρέπει να υποστηρίξουμε εκείνους ε, τους δημοκρατικούς, πολιτισμένους Ιρανούς, να συνεργαστούμε μαζί τους για να διασφαλίσουμε μια ε, αξιοπρεπή ανθρώπινη κυβέρνηση για το καλό του λαού και οι ε, δολοφόνοι να καταδικαστούν. Πάλι άλλο αίτημα παρέμβασης δεν έχουμε. Οπότε, ε, κύριε Επίτροπε, εξ ονόμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχετε το λόγο. <clears throat> Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί από κοντά την περίπτωση Ροξάνα Σαβέρη, συμπληρωμένη και τη προετοιμασία για την διαδικασία τη εξέτασης τη έφεση που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανησυχεί για την υγεία της κυρίας Σαμπέρη εξαιτία τη πρόσφατη απεργίας πείνα. Σήμερα με τον ε, πατέρα της ξεκίνησε την απεργία πίνας μετά την καταδίκη της για υποτιθέμενη κατασκοπιά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η δίκη της κυρίας Σαμπέρη έγινε καταρχήν και κλεισμένο των θυρών και δεν, και δεν ικανοποιεί τι ελάχιστε απαιτήσει για μια δίκαιη και διαφανή δίκη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει πλήρω την δήλωση τη Τσεχική Προεδρία για την περίπτωση Σαμπέρι με ημερομηνία 22 Απριλίου 2009. Ελπίζουμε ότι η Ιρανική δικαιοσύνη θα εξασφαλίσει δίκαιη και διαφανή δίκη σε δεύτερο βαθμό, σχετικά με την έφεση της κυρία ε, Σαμπέρη και θα, ότι θα παράσχει όλες τις εγγυήσει που προβλέπονται βάσει της Ιρανικής νομοθεσίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την βαθιά της ανησυχία για την συνεχή επιδείνωση της κατάστασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών στο Ιράν. Η πρόσφατη εκτέλεση της Νταράμπη, την Πρωτομαγιά, για αδίκημα το οποίο υποτίθεται ότι είχε διαπράξει όταν ήταν ανήλικη, αποτελεί μια ακόμη επιβεβαίωση της απαραδείκτης αυτής κατάστασης. Συνεφώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσίευσε ανακοίνωση με την οποία καταδίκαζε την εκτέλεση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατ' επανάληψη κάλεσε και συνεχίζει να καλεί τις Ιρανικές αρχές να δείξουν το σεβασμό τους για τις διεθνείς τους δεσμεύσεις σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου και μεταξύ αυτών αυτές που απορρέουν από τις διεθνείς συμβάσεις και την διακήρυξη, την διεθνή διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η βελτίωση της κατάστασης ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν είναι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεμελιώδης προϋπόθεση για να μπορέσει να διευρύνει τον πολιτικό διάλογο και την συνεργασία με το Ιράν το προσεχές μέλλον. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, η συζήτηση έληξε. Η ψηφοφορία θα γίνει μετά τη λήξη του συνόλου των συζητήσεων. Και τώρα ερχόμαστε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που προβλέπει έξι προτάσεις ψηφίσματος σχετικά με την Μαγαδασκάρη. Θα ξεκινήσουμε δίνοντας το λόγο στους συντάκτες. Για, για τρία λεπτά το λόγο θα πάρει ο κύριος Ιρίχο Αμεργάνα